τα πρακτικά εγκρίνονται. Ο κύριος Δήμητας Στογιάννοφ έκανε μια πρόταση από 8 Νοεμβρίου 2011 για την ασυλία. Αυτή η πρόταση έχει αποσυρθεί, έχει ληφθεί υπόψη και ε, διαδικασία. Από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, της ομάδας της Αριστεράς και